να αναφέρω το θάνατο ενός συναδέλφου την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μάρκο Πανέλα, ε, επί σειρά τον ε, συναδελφός μας, ε, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί σειρά ετών και εγώ είχα την τιμή προσωπικά να το γνωρίζω. Κυρίε και κύριοι, τον γνώρισα ως έναν ξεχωριστό πραγματικά άνθρωπο με μεγάλο πάθος ε, για την υποστήριξη των ε, πολιτικών δικαιωμάτων, του πλουραλισμού στην κοινωνία μας. Αποτέλεσε ε, πολέμιο της ανατικής καταδίκης, υπέρμαχο των δικαιωμάτων των φυλακισμένων, υπέρμαχο των δικαιωμάτων των ομοφιλόφιλων, της ισότητας των δύο φύλων, όπως πολλοί από τους συναδέλφους μου ε, γνώρισα τον ε, Μάρκο Πανέλα ως ένα ε, Ευρωπαίο υψηλού κύρους και την συμβολή του διευρύνθηκε και επεκτάθηκε πέρα από τα σύνορα της πατρίδας τους και της ομάδας του. Ο κύριος Πανέλα από πολλές απόψεις ήταν ένας πολιτικός πρωτοπόρος και το κριτικό του πνεύμα σε διάφορες περιστάσεις προκάλεσε αμφιλεγόμενες και ακαθώσεις συζητήσεις στην Ευρώπη, στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες και η Ευρώπη χάνει στο πρόσωπο του Μαρκο Πανέλα έναν ε, ένθερμο υποστρεκτή της. Ε, μεταξύ ημών έχουμε σήμερα πολλούς από τους πρώην ε, βοηθούς του και υπαλλήλου του, πολλοί φίλοι του, πολλοί από αυτούς θα συνεχίσουν το έργο τους. Τους κρατίζουμε όλος ιδιαίτερος και εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα θέλαμε να συλληπιθούμε την οικογένεια του κυρίου Πανέλα, δηλαδή, την γυναίκα του και του συνοδοιπόρους του. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα διακόψουμε την σύνοδο